ομάδες. Και τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου, τις τέσσερις μέρες δηλαδή της Συνόδου, το τελικό σχέδιο της ημερήσια διάταξης που υιοθετήθηκε από την διάσκεψη των Προέδρων στις 20, 20 Ιανουαρίου σύμφωνα με τον κανόνα 137 έχει ήδη ε, κοινοποιηθεί στα μέλη. Δεν υπάρχουν αλλαγές για τη Δευτέρα για την ημερήσια διάταξη λοιπόν της Δευτέρας έχει ως ε, αναγράφεται στην ημερήσια σας διάταξη. Για την Τρίτη οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι ζήτησαν για την Τρίτη τη συμπερίληψη μια δήλωση από τον Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή, την είπατε εκπρόσωπο τη Ένωση για τι Εξωτερικέ Υποθέσει και την Πολιτική Ασφάλεια, μια δήλωση για το κράτο δικαίου στην Ρωσία. Θα ήθελαν αυτό να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη τη Τρίτη το πρωί. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Χάρμ, ώστε να κάνει επισήμως το αίτημα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αφενός δεδομένων και των εμπειριών μας με την περίπτωση Χοντοκόφσκι θα πρέπει κατεπηγόντως να συζητήσουμε τι γίνεται με το κράτος δικαίου στη Ρωσία. Αλλά νομίζω ότι εν ώψη και των εκλογών στη Δούμα το φθινόπωρο έχουμε βάσιμους λόγους για να ασχοληθούμε με την κατάσταση της μεγάλης αυτής ε, χώρας στα ανατολικά της Υπήρου. Νομίζω ότι σήμερα είναι επίκαιρο όλοι να ασχοληθούμε και να κοιτάξουμε κατά πόσο ε, δεσμευόμαστε στην, ε, στις γειτονικές μας χώρες για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των πολιτικών δικαιωμάτων και πολλοί έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση αν για τα θέματα της Τινησίας, της Αιγύπτου συζητήσαμε τα απαραίτητα ζητήματα. Δεν θέλω μια τέτοια αμέλεια να επιτραπεί στα ανατολικά της Υπήρου μας. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ και απευθύνω έκκληση να συζητήσουμε αύριο το θέμα του κράτους δικαίου στην Ρωσία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φερχόφστατ θα ήθελε να υποστηρίξει αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να υποστηρίξω το αίτημα της Ρεμπέκα Χάρμς και θα πρέπει επίσης να σας πω ότι αφού του διατυπώσαμε το αίτημα αυτό στη διάσκεψη των Προέδρων και τώρα εδώ στην Ολομέλεια της Συνόδου λαμβάνουμε όλο ένα και μεγαλύτερη πίεση, ασκείται μάλλον όλο ένα και ε, μεγαλύτερη πίεση από την ρωσική πλευρά για να μην ε, συζητηθεί το θέμα και η κυρία Λόγελα. Επίσης την περασμένη εβδομάδα ε, που διοργάνωνε σεμινάριο για το κράτος δικαίου στη Ρωσία ε, δέχθη πίεση για να μην συζητηθεί το θέμα του κράτους δικαίου για τη Ρωσία αλλά δεν είναι θέμα των Ρώσων να αποφασίσουν την ημερήσια διάταξή μας. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε για την ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου. Θέλει κάποιος να μιλήσει κατά. Κύριε Σεβερίν, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ως μόνιμος εισηγητής για τις σχέσεις με τη Ρωσία, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ήδη ξεκινήσαμε μια πολύ εις βάθος διαδικασία ώστε να ασχοληθούμε με όλα τα σοβαρά ζητήματα που είναι σημαντικά για τη σχέση μας με τη Ρωσία. Ήδη είχαμε μια ακρόαση με τον εκπρόσωπο, τη, την εκπρόσωπο της εξωτερικής υπηρεσίας και εκπρόσωπο της ρωσικής κυβέρνησης. Στις 2 Μαρτίου οργανώνεται μια άλλη ακρόαση με εμπειρογνώμονες που θα εξετάσουν όλες τις σημαντικές πτυχές των σχέσεών μας με τη Ρωσία. Τη δεύτερη δεβδομάδα του Μαρτίου προγραμματίζεται ένα κείμενο που συμπεριλαμβάνει σύσταση για το οποίο θα τεθεί υποσυζήτηση και θα είναι ανοιχτό σε τροπολογίες και που θα καταλήξει σε συζήτηση στην Ολομέλεια με τη συμμετοχή της ΥΠΑ της εκπροσώπου που από όσο γνωρίζουμε δεν είναι διαθέσιμη για αυτή την εβδομάδα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως χωρίς να παραμελούμε ή να αρνούμεθα τη σημασία του θέματος θα ήταν πολύ καλύτερο να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και να φτάσει στην ολοκληρωσή της με τρόπο ώστε να έχουμε μια τεκμηριωμένη συζήτηση που θα μας επιτρέψει να είμαστε και πιο αξιόπιστοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ψηφίσουμε. Έχετε διαδικαστικό, μάλιστα. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Την περασμένη εβδομάδα, στην διάσκεψη των Προέδρων, είπαμε ότι θα γίνει συζήτηση για τη Ρωσία τον Μάρτιο, γιατί η κυρία Άστον θα είναι παρούσα. Και έπειτα Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των Προέδρων είπαμε πρέπει να γίνει συζήτηση για τη Ρωσία γιατί ο κύριος Πούτιν έρχεται να κάνει μια επίσκεψη στην Κομισιόν, στον κύριο Μπαρόζο. Οι πληροφορίες που έλαβα σήμερα το απόγευμα είναι ότι ο κύριος Πούτιν δεν θα έρθει, δεν θα επισκεφθεί την Κομισιόν. Έχετε εσείς κάποια ενημέρωση, πληροφορίες ή τίποτα το ζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα γιατί θα ερχόταν ο κύριος Πούτιν. Γιατί διαφορετικά ούτως ή άλλως προβλέπεται συζήτηση για τη Ρωσία με ψήφισμα για το Μάρτιο. Ήταν διαδικαστικό, ναι, το καταλαβαίνω. Αν θέλετε κι εσείς σε κάποιο διαδικαστικό να κάνετε, όχι. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε τώρα. Τώρα θα ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης των Πρασίνων και Φιλελευθέρων. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την πρόταση αυτή. Σοβάνιε. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η πρόταση. Εγκρίνεται η πρόταση, κυρίες και κύριοι. Η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου για το κράτος δικαίου στην Ρωσία θα συμπεριληφθεί στην αυριανή ημερήσια διάταξη ως τρίτο σημείο. Τρίτο σημείο λοιπόν για την πρωινή ημερήσια διάταξη της Τρίτης. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 10 το πρωί αύριο. και η προθεσμία για τα κοινά ψηφίσματα ή τις κοινέ προτάσεις ψηφισμάτων είναι την ε, Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί. Και για την, είναι τελική επίσης ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Και η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, έχω ακόμα ένα αίτημα σε σχέση με την ημερήσια διάταξη της Τρίτης. Ε, το ΕΛΚ έχει ζητήσει τη συμπερίληψη μιας δήλωσης από πλευράς της Κομισιόν για την κατάσταση στη Λαμπεντούζα. Θα ακούσουμε τον κύριο Μάριο Μάουρο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, σωστά θυμήσατε, είμαστε ε, μπροστά σε εποχιακά φαινόμενα τα οποία καθορίζουν μια έκτακτη αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Βεβαίω, αυτή τη στιγμή η Λαμπαντούζα ε, δέχεται, έχει κατακλειστεί από αυτή την ε, εισρωή μεταναστών, αλλά καλείται φυσικά ολόκληρη η Ευρώπη για τη διαχείριση ε, των αλλαγών που περνά ολόκληρο το Μαγκρέμπ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Κομισιό να λάβει το λόγο και να απαντήσει όχι μόνο στα ανθρωπιστικά ζητήματα, αλλά και στα πιο βαθιά στρατηγικά ζητήματα που πρέπει να μας οδηγήσουν να θεωρήσουμε την πολιτική μας σε σχέση με τη Μεσόγειο. Ζητούμε λοιπόν την Τρίτη να γίνει μια χωριστή συζήτηση το απόγευμα με την Επίτροπο Μάλνστρομ και να περιοριστεί ο χρόνος της, των ερωτήσεων προς την Επιτροπή κατά μισή ώρα δεδομένη σημασία του ζητήματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Σούλτ θα μιλήσει υπέρ του αιτήματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ως σοσιαλδημοκράτες έχουμε και εμείς να υποβάλουμε την ίδια, το ίδιο αίτημα. Ωστόσο, θα ήθελα προς τον συνάδελφο Μαωρό και προς την Βουλή να προτείνω να είμαστε κάπως πιο συγκεκριμένοι. Γιατί είναι τεράστια εισρωή η Ιταλία, όπως και κάθε άλλη χώρα της Μεσογείου, έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ και δεν μπορεί να επιλύσει μόνο το πρόβλημα. Και σίγουρα δεν θα είναι μόνο η Ιταλία το, η μοναδική χώρα που θα αντιμετωπίσει τέτοιο τεράστιο κύμα μεταναστών. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και η Μάλτα και η Ελλάδα και η Ισπανία σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωπε με τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να απευθύνουμε την εξή έκκληση, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στην ε, διατύπωση του αιτήματο μα, δηλαδή μέτρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη τη Ιταλία και άλλων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πλήττονται κατά την αντιμετώπιση τη ροή μεταναστών. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κανείς να μιλήσει κατά αυτή τη πρόταση. Nobody. this. Ωραία. Θα προσχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Όσοι είναι υπέρ, τι θέλετε να μιλήσετε κατά. Κατά, ποιος είναι κατά. Α, συνάδελφοι. Ψηφίζουμε τώρα για την πρόταση του Μάριο Μάουρο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, σας ευχαριστώ. Διαδικαστικό. Εγκρίνεται. Μισό λεπτό παρακαλώ. Και το σημείο αυτό θα συμπεριληφθεί ως δεύτερο σημείο στην απογευματινή ημερήσια διάταξη της Τρίτης. 6.30 με 7.30 το απόγευμα. Είναι το δεύτερο σημείο στην απογευματινή ημερήσια διάταξη της Τρίτης και η ώρα των ερωτήσεων θα μετακινηθεί. Συγγνώμη, κατά μισή ώρα, 6,5 με 7,5. Πάμε τώρα στον τίτλο της συζήτησης αυτής. Κάποιος θέλει να μιλήσει σε σχέση με τον τίτλο της συζήτησης. President, I want to Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να υποστηρίσω την πρόταση του κυρίου Σούλτ. Γιατί είναι πολύ ευρύτερο το πρόβλημα από την Λαμπεντούζα. Έχουμε 5 χιλιόμετρα από το Μαρόκο μέχρι τη Συρία. Και κάθε χιλιόμετρο παρουσιάζει αυξανόμενο ανθρωπιστικό κίνδυνο. Δεν είναι θέμα να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει την Ιταλική κυβέρνηση, αλλά αν είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε ω ήπειρος για να αντιμετωπίσουμε έναν ε, ε, κίνδυνο για όλους. Έχετε δίκιο συνάδελφοι, γι' αυτό ψηφίσαμε και θα το συζητήσουμε όπως, ε, όπως φάνηκε. Θα το συζητηθεί το θέμα, άρα όλα πάνε καλά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να μιλήσουμε για τον τίτλο αυτής της συζήτησης. Η ομάδα των σοσιαλιστών προτείνει να είναι ευρωπαϊκά, ε, μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ιταλίας σε σύνδεση με, τη, ε, με τις μεταναστευτικές ροές, το μεταναστευτικό κύμα. Ο πρόεδρος Σουλτς θέλει να το τροποποιήσει αυτό νομίζω. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να διευκρινίσω και πάλι. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κάνει δήλωση για καταπήγοντα άμεσα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ιταλίας και άλλων χωρών που πλήττονται κατά την αντιμετώπιση της εισρωής του κύματος ε, μεταναστών. Ωραία. Έγινε κατανοητό. Ο τίτλος λοιπόν που προτείνεται είναι μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη της Ιταλίας και άλλων χωρών που πλήττονται από ασυνήθιστα μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Ποιο είναι υπέρ του τίτλου αυτού παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν ο τίτλος. Με μεγάλη πλειοψηφία η οποία στήριξε αυτή την απόφαση. Σε ό,τι αφορά την Τετάρτη δεν έχουμε προτάσεις για τροποποίηση της μερίσιας διάταξης, περνώ στην Πέμπτη η ομάδα της Ευρώπης της Ελευθερίας και Δημοκρατίας έχει ζητήσει να συμπεριληφθεί προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης στην περίπτωση του Τζούλιαν Ασάντζ. Ποιο θα μιλήσει υπέρ του αιτήματο αυτού, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωτή. Η προφορική αυτή ερώτηση δεν αφορά το κατά πόσον είναι ένοχο ή αθώο ε, ο κύριο Ασάντ σε ό,τι αφορά τι κατηγορίε βιασμού για την ε, Σουηδία. Έχει να κάνει με τη χρήση ή κατάχρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματο ε, Σύλληψη για πολιτικού λόγου. Με το Ευρωπαϊκό Εντάλμα Σύλληψη κάθε πολίτη μπορεί να παραδοθεί χωρί να υπάρξει ε, η, χρήση του πρίμα φάκιες αυτού του νομικού ε, επιχειρήματος και εκεί υπάρχουν ε, πάρα πολλά μεγάλα περιθώρια χρήσης και κατάχρησης κατά πολιτικών αντιφρονούντων. Για τα υποτιθέμενα λοιπόν αξιόπινα, αξιόπινες πράξεις του διασμού του Τζούλιαν Ασάντς πρόκειται ή μήπως ε, για κάποιους άλλους ε, λόγους ε, και που έχουν να κάνουν με τις ΗΠΑ. Πρέπει να κατανοήσουμε τους λόγους για να αποφασίσουμε κατά πόσον υπάρχει κακή χρήση, κατάχρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Νομίζω ότι πρέπει όλο το πολιτικό φάσμα στο Κοινοβούλιο να το συζητήσει αυτό το θέμα. Σας ζητώ λοιπόν να υπερψηφίσετε το έτοιμά μας. Ο Πρόεδρος σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα ήθελε να μιλήσει υπέρ αυτού του αιτήματο. Κυρία Χέρτσοκ, υπέρ. Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω το 2004 ένας Ιρλανδός ε, υπάλληλο προκάλεσε ένα θαντιφόρο ατύχημα στην Ουγγαρία και την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία ε, λάβαμε τη απόφαση των Ιρλανδικών ε, αρχών ότι μπορεί να ε, επιστραφεί ο άνθρωπος αυτός στο δικαστήριο της Ουγγαρίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία και θα πρέπει να ενισχυθεί. Δ'άλλως τα θύματα θα πρέπει να περιμένουν χρόνια ολόκληρα, όχι μόνο άμα σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Άρα είμαστε σαφώς υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να είμαστε λίγο ήσυχοι στην αίθουσα. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να μιλήσει κατά αυτού του αιτήματο. Είστε κατά. Κατά. Yes, please. Παρακαλώ. Πρόεδρε. Ένα δικαστικό να διευκρινίσω. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση, αν μπορούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουμε μία ε, συζήτηση επί της αρχής για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά τώρα κατά πόσο μπορούμε να τη συνδέσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο με μία διαδικασία, με μία εκδίκαση η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δεν το ξέρω αυτό. Θα ήθελα να το συνδέσω και με άλλες περιπτώσεις, αν ε, είναι δυνατόν, αλλά θα ήθελα να μην καταστήσουμε αυτή την υπόθεση η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχει εκδικαστεί ε, αντικείμενο της συζήτησής μας. Σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Έχουμε λοιπόν αυτό το αίτημα από την ομάδα της Ευρώπης ε, της Ελευθερίας και Δημοκρατίας, οποίοι θα ήθελαν προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης ε, για την περίπτωση Τζούλιαν Ασάντς. Να συμπεριληφθεί αυτή η ερώτηση. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Σας ευχαριστώ. Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα. Ως εκ τούτου εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στις εργασίες της Συνόδου. Παρακαλώ να υπάρξει ησυχία και όποιοι θέλουν να αποχωρήσουν να το πράξουν ησύχως. Αλλιώς να παραμείνουν παρακαλώ. Dear colleagues, please, one minute. Αγαπητοί συνάδελφοι,